το λόγο. Παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, δυστυχώς πρέπει να σας ενημερώσω ότι μόλις μάθαμε ότι το γενικό το στρατηγείο των Ηνωμένων Εθνών για την βοήθεια των, που προσφέρει βοήθεια στους πρόσφυγες στη Γάζα μόλις βομβαρδίστηκε από τους Ισραηλινούς και ως εκ τούτου ο ΙΕ αποφάσισε να σταματήσει πάσα δραστηριότητα. Λόγω και της ψηφοφορίας που επίκειται είναι νομίζω σημαντικό όλοι μας να γνωρίζουμε τι συνέβη. Vielen Dank, Herr Ευχαριστούμε κύριε Βούρτς για αυτή την πληροφορία.